να δώσει περαιτέρω εξήγηση. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τις ε, παρεμβάσεις σας. Σας ενημερώνω πως η συνεδρία θα επαναληφθεί αύριο το πρωί σε 9. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.